εξ ονόματος του Συμβουλίου στην Υπουργό Χένις Πλάσχαρτ. Έχετε το λόγο. Oczywiście e, Λίγα λεπτά διακοπή και μετά ούτως ώστε ε, να μιλήσετε και μετά θα μιλήσει ο Επίτροπος Χάν και μετά θα έχουμε ομιλητές εκ μέρους των πολιτικών ομάδων. Επίσης θα λάβω και εγώ τον λόγο σε αυτή τη συζήτηση. Θα πρέπει να αντικατασταθώ εδώ ως Αντιπρόεδρος και για να μπορέσω να λάβω τον λόγο. Ε, η κυρία Υπουργός Χενής Πλασέρτ έχει τον λόγο. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να επαναλάβω την δέσμευση ε, του Συμβουλίου για την διαδικασία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Η κατάσταση είναι κρίσιμη στην χώρα και μας ανησυχεί. Το 2015 η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας είχε από τις σοβαρέτερες πολιτικές κρίσεις και έχουμε την οπισθοχώρηση της ελευθερίας έκφρασης και της ε, ελευθερίας και ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και διάβρωση των ε, πολιτικών θεσμών. Θα πρέπει να ξεπεραστεί η κρίση και ε, τα σχόλια αυτά να είναι χρήσιμα. Η συμφωνία μεταξύ τον Ιούλιο μεταξύ των πολιτικών κομμάτων και οι προτεραιότητες της Κομισιόν δίνουν το υπόδειγμα για το τι πρέπει να γίνει. Έχουμε σημειώσει την απόφαση για, ε, για τις 5 Ιουνίου της αναβολής των εκλογών, ώστε να υπάρξουν οι ε, συνθήκες ε, οι κατάλληλες θα είναι ουσιαστικό για όλους τους πολιτικούς φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους και να λάβουν μέτρα ακόμα και ε, την μεταρρύθμιση για τα μέσα για τις εκλογές. Θα πρέπει να υπάρξει διάλογος χωρίς αποκλεισμού στην χώρα. Είναι κάτι το κρίσιμο για την πρόοδο. Και η οργάνωση ε, αξιόπιστων εκλογών όπου όλα τα άτομα και τα κόμματα θα συμμετάσχουν θα είναι ένα πρώτο μεγάλο βήμα για να τέθει τέρμα στην πολιτική κρίση. Παρακολουθούμε ε, εκ του ε, με, το Γραφείο για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και συνιστώ στενή συνεργασία ανάμεσα με την Ηνωμένα Έθνη ούτως ώστε να βγει η χώρα από την κρίση και θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα τις προσπάθειες του Επιτρόπου Χάν, τον ευχαριστώ και των τριών μελών των τριών Ευρωβουλευτών Φάιφερ, Χάλο και Κούκα που ασχολήθηκαν με το θέμα. Σας ευχαριστώ πολύ θα έχουν ασχοληθεί με τα θέματα κράτους δικαίου, δημόσιας δίκησης, προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, την καταπολέμηση της διαφθοράς που παραμένει ε, μεγάλο πρόβλημα ούτω ώστε να οδεύσει προς την Ευρωπαϊκή Ένωση χώρα. Επαναλαμβάνουμε την σημασία ανεξαρτήτων ερευνών για όλες τις καταγγελίες που έχουν γίνει. Ο ειδικό εισαγγελέα και η Επιτροπή Κοινοβουλευτική, η Εξεταστική θα πρέπει να υποστηριχθούν και θα ήθελα να επαναλάβω την έκκληση ε, του Συμβουλίου ε, σχετικά με τα γεγονότα στο Κουμάνοβο που θα πρέπει να εξεταστούν ε, με σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με ε, την, το προσφυγικό. Θα ήθελα να συγχαρώ την Δημοκρατία ε, για τις προσπάθειες που κατέβαλε πέρσι για το προσφυγικό εδώ ε, και μερικές εβδομάδες, μερικές αποφάσεις μονομερείς λήφθηκαν στην οδό των Δυτικών Βαλκανίων το Συμβούλιο στις 18 ε, Φεβρουαρίου ήταν ε, σαφές ότι μόνο συμπεφωνημένη δράση μπορεί να αντιμετωπίσει την πρόκληση με κατάλληλο τρόπο. Δεν υπάρχει εναλλακτική λύση ε, άλλη από μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή λύση και θα πρέπει η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ως γειτονική χώρα και υποψήφια χώρα να παίξει το ρόλο της σε αυτή τη διαδικασία. Ευρωπαϊκή Ένωση παρέχει υποστήριξη σε αυτήν την δημοκρατία ούτως ώστε να ενισχύσει τους έλεγχους στα σύνορα και να βελτιωθεί η διαδικασία του ασύλου ε, ε, ε, και γίνονται προσπάθειες σε διμερές επίπεδο. Οι καλές χώρες, οι καλές σχέσεις γειτονίας θα επιτρέψουν λύσεις υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών και είναι σημαντικές για την σταθερότητα. Η ενταξιακή διαδικασία της χώρας βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή. Η Επιτροπή είναι διατεθειμένη ε, να παρατείνει τις ε, συστάσεις για ανοιχτές διαπραγματεύσεις, αλλά υπάρχουν ε, συνθήκες, όροι να εφαρμοστεί η Συμφωνία η Πολιτική Ιουνίου-Ιουλίου και να γίνει πρόοδος στην εφαρμογή των ε, μεταρρυθμίσεων που είναι επίγουσες προτεραιότητες. Ανεφερόμεθα ε, θα ασχοληθούμε μετά τις εκλογές με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Νομίζω τώρα ότι οι πολιτικοί ηγέτες έχουν την ευθύνη να λάβουν τα απαιτούμενα ε, μέτρα ούτως ώστε ε, να μπει σε σωστή τροχιά η χώρα. Ευχαριστώ πολύ και τώρα εκ μέρους της Επιτροπής ο Επίτροπος Ιωάννης Χάν. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θέλω να ευχαριστήσω την ε, Πρόεδρο του Συμβουλίου για τα καλά της λόγια αλλά θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάγκελ, τον κύριο Κούκαν, τον κύριο Χάουιτ για την ε, αδιάκοπη προσπάθειά της να βοηθηθεί η χώρα αυτή και να διευκολυνθούν οι προσπάθειες μαζί με την Κομισιόν οι προσπάθειες για την επίτευξη μιας πολιτικής λύσης από πέρσι το καλοκαίρι. Είναι κεφαλαιόδες να βοηθήσουμε την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αντιμετωπίσει τις ε, μεγάλες πολιτικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει τώρα και να τήρηθει η πολιτική συμφωνία που έχει επιτευχθεί ζωντανή και τους επερχόμενους μήνες. Οι τρεις βουλευτές πήγανε στην ε, Ποδογομού πριν από ένα μήνα περίπου μετά από την ε, επιστολή των, του Πρεσβευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παρουσίασε την ε, κοινή θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι οι συνθήκες για τη διενέργεια εκλογών στις 24 Απριλίου δεν πληρούντο. Μαζί με την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι τρεις συνάδελφοί σας επέτυχαν μια συμφωνία των πολιτικών δυνάμεων για να αναβληθούν οι πρόορες εκλογές μέχρι τις 5 Ιουνίου του έτους αυτού και θέλω να τονίσω πόσο σημαντικό είναι αυτό ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έπαιξε ένα σημαντικό ρόλο για να βοηθήσει να προχωρήσει σωστά η δημοκρατική διαδικασία και θέλω να εκφράσω την επιθυμία και την ευχή ότι θα είναι δυνατό να είμαστε παρόντες με παρατηρητές την εποχή των εκλογών. Θέλω να τονίσω επίσης ότι αυτό είναι μια ευκαιρία να ευχαριστήσω τον Ιβο Βάγγλ, τον εισηγητή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για το ψήφισμα το οποίο παρουσιάζεται σήμερα ενώπιόν σας για έγκριση. Είναι εξισορροπημένο και συνάδει με τα κύρια πορίσματα της έκθεσής μας το 2015 για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Όπως ξέρετε ήταν μια δύσκολη περίοδος αυτή που καλύπτεται από την έκθεση, αλλά είμαστε πεπισμένοι ότι η έκθεσή μας έχει επιτύχει τη σωστή ισορροπία. Από τη μία πλευρά αναγνωρίζουμε ότι υπήρξε ένα σημαντικό επίπεδο προετοιμασίας της χώρας αυτής, έχει μια λειτουργούσα οικονομία της αγοράς, έχει σχετικά καλή ε, προσαρμογή στο ευρωπαϊκό κεκτημένο. Αυτό σημαίνει ότι οι σωστοί νόμοι και στρατηγικές είναι, είναι στη θέση τους, αλλά το βασικό πρόβλημα στη χώρα αυτή είναι η εφαρμογή και η παρακολούθηση αυτής της ε, εφαρμογής της νομοθεσίας. Η χώρα αυτή έχει αντιμετωπίσει μια από τις πιο σοβαρές πολιτικές κρίσεις εδώ και πολλά χρόνια μποϊκοταρίστηκε από το κόμμα της αντιπολίτευσης για πάνω από ένα χρόνο το κοινοβούλιο της ε, χώρας αυτής και η κατάσταση επιδεινώθηκε με τη δημοσίευση υποκλαπισών συνομιλιών που καταδεικνύει ότι έχει υπάρξει υψηλού επίπεδου διαφθορά και η υπονόμευση του δικαστικού συστήματος. Για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε αυτή την κρίση, ακολουθήσαμε μια διτή προσέγγιση. Πρώτα απ' όλα την πολιτική συμφωνία μεταξύ των κομμάτων που επετεύχθη από τους τέσσερις ηγέτες των μεγάλων πολιτικών κομμάτων πέρσι το καλοκαίρι και αυτό ήταν ένα αποφασιστικό βήμα προς το εμπρό. Μερικές από τις δεσμεύσεις έχουν υλοποιηθεί μέσα στην προβλεπόμενη ε, μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα γύρισε το κόμμα της αντιπολίτευσης στο Κοινοβούλιο και ένας ειδικό εισαγγελέα διορίστηκε το φθινοπροπέση. Αλλά άλλες δεσμεύσεις δεν έχουν τηρηθεί και χρειάζεται η ενεργή δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να προωθηθούν. Μαζί με την πολιτική συμφωνία του Ιουνίου εμείς παρουσιάσαμε ένα σύνολο <clears throat> προτεραιοτήτων, κατεπηγουσών προτεραιοτήτων ε, μεταρρύθμισης για να αντιμετωπιστούν τα θέματα του κράτους δικαίου και πάλι όλα αυτά είναι πάρα πολύ κεφαλαίωδη. Στην έκθεσή μας τονίσαμε ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να συνεχίσει τη σύστασή της για, την, για το άνοιγμα διαπραγματεύσεων με τη χώρα αυτή με την προϋπόθεση ότι θα συνεχιστεί να εφαρμόζεται η συμφωνία του Ιουνίου-Ιουλίου του 2015 και την υλοποίηση των προτεραιοτήτων που έχουν αναφερθεί. Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τα θέματα αυτά και θα σας παρουσιάσουμε μια έκθεση εν ευθέτω χρόνο. Όπως πολύ, πολύ καλά αναφέρει το ψήφισμα του Κοινοβουλίου, η Ιντερεθνική η κατάσταση μεταξύ των εθνοτήτων στην χώρα αυτή παραμένει τεταμένη. Θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα αυτά τα θέματα μεταξύ εθνοτήτων και να δημιουργηθεί και πάλι εμπιστοσύνη μεταξύ των διαφορετικών εθνοτικών κοινοτήτων και πρέπει να συνεχιστεί η αναθεώρηση της Συμφωνίας της Αχρίδας. Είναι απαραίτητες αυτές οι καλές σχέσεις μέσα στη χώρα και σε εξωτερικό επίπεδο η επίλυση του θέματος του ονόματος είναι και αυτή μια προτεραιότητα και οι χώρες αυτές που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του <clears throat> προσφυγικού ρεύματος παίζουν σημαντικό ρόλο και η Κομισιόν είναι προσιλωμένη στο να συνεχίσει τη βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Για όλους αυτούς τους λόγους προσβλέπω στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε στον κύκλο των εισηγητών εκ μέρους των πολιτικών ομάδων στη συζήτηση για την έκθεση προόδου για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας για το 2015. Το λόγο έχει για δύο λεπτά για την Συμμαχία των Φιλελευθέρων και Δημοκρατών ο κύριος Βάγκλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Χένις Πλασάρτ, κύριε Πίτροπε Χάνα. Καταρχάς, θα πρέπει να πω ότι οφείλω να σας ευχαριστήσω για τα πολύ θετικά λόγια τα οποία είπατε όσον αφορά τη συνεργασία που είχαμε. Και πρέπει να πω επίσης ότι ε, Είχα και εγώ την ίδια ευχαρίστηση κάθε φορά που συνεργαζόμουν μαζί σας. Εγκρίνουμε αυτή τη στιγμή από κοινού μία, ένα ψήφισμα για την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, μόλον ότι είχαμε 300 τροπολογίες. Θεωρώ όμω ότι ε, καθυστερήσαμε πάρα πολύ με την έκθεση αυτή. Καθυστερήσαμε όμως πάρα πολύ να δεχθούμε και την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ανάμεσα στις χώρες αυτές που πρέπει να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια χώρα που πλήττεται πάρα πολύ από την προσφυγική κρίση αυτή τη στιγμή. Στις 5 Ιουνίου θα γίνουν πρόορες εκλογές στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και κατά αυτόν τον τρόπο θα τεθεί τέλος στην πολιτική κρίση. Αν ακολουθηθούν δημοκρατικά πρότυπα στις βουλευτικές αυτές εκλογές, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα είναι σε θέση να εγκρίνουν την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων για προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπό τους ίδιους όρους που προβλέπονται και για τις υπόλοιπε χώρε. Η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας αντιστοιχεί αυτή τη στιγμή και πληρεί το μεγαλύτερο μέρο του κοινοτικού κεκτημένου και δημιουργεί σχέσει καλή γειτονία με τι όμορε τη χώρε και συμβάλλει επικοδομητικά στο να οικοδομηθεί εμπιστοσύνη με τι χώρε εκείνε όπω η Ελλάδα, η Βουλγαρία που έχει ακόμα κάποια κρεμή ζητήματα. Στο ψήφισμα αυτό, όπω και στη σχετική έκθεση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναφερόμαστε σε κάποια ζητήματα τα οποία έχουν προκύψει ιδίως όσον αφορά τις υποκλοπές των συνδιαλέξεων. Είπαμε ότι ε, θα πρέπει να ισχύσει η συμφωνία της Πρίστινας προκειμένου να έχουμε πραγματικά ένα γραφείο του ειδικού εισαγγελέα ο οποίος να μπορεί να λειτουργεί πλήρως. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο θα καταφέρουμε να έχουμε ένα δημοκρατικό καθεστώς και ανάλογες μεταρρυθμίσεις πρέπει να γίνουν προκειμένου να έχουμε πλέον μια ε, θετική ε, συνύπαρξη ανάμεσα στα διάφορα πολιτικά κόμματα της χώρας. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να έχουμε και τη συμβολή της διαμεσολάβησης τόσο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου όσο και εκπροσώπων των ΗΠΑ. Κυρίες και κύριοι, θα πρέπει η πρώην Κωνσταντική Δημοκρατία της Μακεδονίας να αρχίσει να κινείται στην ευρωατλαντική της πορεία. Και η δική μου ομάδα υποστηρίζει αυτή την προοπτική. Λυπάμαι που δώσαμε ελάχιστο χρόνο στην εξέταση της έκθεσης αυτής. Έχετε μια μπλε κάρτα από την κυρία Βόζεμπεργκ. Δέχεστε αυτή την μπλε κάρτα, κύριε Βάιγκελ. Oui, madame Βόζεμπεργκ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, άκουσα με προσοχή τις ε, τοποθετήσεις σας σε σχέση με τη Φύρομ. Γνωρίζετε ότι αυτή τη στιγμή έχει χτίσει φράκτες, έχει ρίξει δακρυγόνα, έχουν συσσωρευτεί άνθρωποι απελπισμένοι, οι οποίοι βρίσκονται σε επίπεδο ανθρωπιστικής κρίσης. Κατά την άποψή σας, η στάση αυτή της Φύρομ απέναντι σε αυτό το πολύ σημαντικό ευρωπαϊκό πρόβλημα θα πρέπει να ληφθεί υπόψη εν ώψη των ενταξιακών συνομιλιών της προς την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Για να απαντήσετε. Κοιτάξτε, δεν μπόρεσα να παρακολουθήσω πολύ καλά την ε, διερμηνία και δεν μπόρεσα να καταλάβω πάρα πολύ καλά την ουσία του ερωτήματός σας. Ωστόσο, να φανταστώ λίγο τι μπορεί να ρωτήσατε. Προφανώς το πρόβλημα αυτό είναι τεράστιο για μια μικρή χώρα, η οποία καλείται αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει ένα τόσο τεράστιο πρόβλημα στα σύνορά της. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και γενικότερα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στηρίξει την Μακεδονία, λέει για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα στα σύνορά της. Αν αυτό ήταν το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για την ομάδα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για ένα λεπτό, ο κύριος Κέλαμ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κυρία Υπουργέ, κύριε Επίτροπε, θα ήθελα να ευχαριστώ τον εισηγητή Βάγγελ για την καλή προσέγγιση και για την, ε, την προσπάθεια να αντιμετωπίσει ένα περίπλοκο θέμα. Η Μακεδονία υπήρξε υποψήφια εδώ και δέκα χρόνια, όπως και θεωρήθηκε προχωρημένη υποψήφια. Ωστόσο, η έναρξη των διαπραγματεύσεων ε, μπλοκαρίστηκε για χρόνια στο Συμβούλιο. Εδώ σε αυτήν την έκθεση γίνεται λόγος για την ανάγκη σταθεροποίησης και ε, καλής συνεργασία με τους διάφορους φορείς, διότι ο διάλογος, η αμοιβαίος σεβασμός και η τήρηση των βασικών αρχών όπως της ελευθερίας του τύπου είναι απαραίτητα στοιχεία για να υπάρξει κράτος δικαίου. Βεβαίως, ε, δεν λειτουργεί καλά η δημοκρατία όπως το βλέπουμε με τις εκλογές και είναι κάτι το επιζήμιο για την χώρα. Οι εκλογές θα είναι σημαντικές για όλους μας και θα ε, πρέπει να τηρηθεί η συμφωνία ε, του Κουμάνοβο. Ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Εγώ υπήρξα εισηγητής και τώρα είμαι σκιώδης εισηγητής και ουσιαστικά διαμεσολαβητής για την χώρα αυτή, αλλά είμαι απόλυτα προσιλωμένος στην προοπτική ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από την πλευρά του, των σοσιαλιστών χαίρομαι πάρα πολύ που μπορέσαμε να ξεπεράσουμε τις κομματικές διαφορές μου και μαζί με το ΕΛΚ και, την, και τους φιλελευθέρους μπορέσαμε να ενθαρρύνουμε τις πολιτικές ομάδες στα Σκόπια να επιλύσουν τις διαφορές τους. Άρα παραμένει ένα πραγματικό ερώτημα. Δεν ξέρουμε ακόμα αν υπάρχει δημοκρατική δέσμευση από τα κόμματα αυτά. Έχουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε ένα σημαντικό ερώτημα. Όπω είπε ο κύριο Χάνη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει τη σύσταση να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσει με την προπόθεση τη πλήρου εφαρμογή τη συμφωνία των κομμάτων που βοηθήσαμε εμεί να επιτύχουμε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον υποστήριξε στα συμπεράσματα του, του Δεκεμβρίου και αύριο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να σταθεί μαζί του και να πει υποστήριξε τη δημοκρατία σας, αλλιώς δεν θα υπάρξει θετική γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν υπήρξε και μια κρίση όταν το κυβερνό κόμμα είπε ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις για τα μέσα ενημέρωσης. Εμείς καταγράψαμε ως μεσολαβητές ότι αυτό δεν ήταν κομμάτι καμία συμφωνίας και χαίρομαι που η Ολλανδική Προεδρία το επανέλαβε σήμερα. Η θέση του Συμβουλίου και της Κομισιόν και που υποστηρίζει τα απόλυτα από το Κοινοβούλιο είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να γίνεται πρόοδος για τις κατεπίγουσες μεταρρυθμίσεις και ο Επίτροπος Χάν μας είπε ότι υπήρχαν, υπήρξαν κάποιες υποχωρήσεις, υπαναχωρήσεις. Ο ειδικό εισαγγελέα λοιπόν για την εγκληματικότητα εναντίον των πολιτικών μας είπε ότι αυτή η ίδια δεν έχει λάβει την πλήρη συνεργασία που θα έπρεπε να έχει από το κρατικό σύστημα Δικαιοσύνη, Πρέπει εμεί να επιμείνουμε αύριο να έχει απόλυτη, ε, απόλυτη αυτονομία και τι απαραίτητε εξουσίε να συνεχίσει την ερευνά τη, Εγώ και η ομάδα μου δεν θα χρησιμοποιήσει το γεγονό ότι η χώρα αυτή βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα τη προσφυγική κρίση για να τη επιτεθούμε. Θέλουμε να έχουμε αλληλεγγύη με τα Σκόπια και χρειάζεται αλληλεγγύη από όλε τι χώρε εάν πρόκειται να προκύψει μια σωστή αντιμετώπιση του προβλήματο αυτού. Αλλά σήμερα πρέπει να στείλουμε ένα στεναρό αλλά και αυστηρό μήνυμα ότι οι πολιτικοί της χώρας αυτής δεν έχουν εκπληρώσει τα υπεσχημένα, αλλά δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτή την υποχρέωση. Αυτό δεν είναι εναντίον του μακεδονικού λαού, αλλά υπέρ του μακεδονικού λαού για τη δημοκρατία της χώρας αυτής και ένα καλύτερο μέλλον και είμαστε σίγουροι θα τους πούμε ότι αυτό θέλουμε και αυτό θέλετε κι εσείς και οι πολιτικοί σας θα πρέπει να δείξουν ότι και αυτοί, αυτοί, το θέλουν επίσης. Ναι. Μπλε κάρτα από την κυρία Σακοράφα κύριε Χάουιτ. Τη δέχεστε? Κυρία Σακοράφα, έχετε 30 δευτερόλεπτα για την ερώτηση. Κύριε Χάουιτ, το ψήφισμα στην αιτιολογική σκέψη G αναφέρει ότι η Επιτροπή, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο συμφωνούν πω η διατήρηση εθνική σύσταση όσον αφορά την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη χώρα εξαρτάται από την πλήρη εφαρμογή τη πολιτική συμφωνία Ιουνίου Ιουνίου-Ιλίου 2015 και την ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή των επιγουσών μεταρρυθμιστικών προτεραιοτήτων. Έχω μια απορία Πού το έχετε δει αυτό και αναφέρομαι σε εσά, κάνω την ερώτηση σε εσά γιατί είναι δική σα αυτή η τροπολογία. Το Συμβούλιο στι 15 Δεκεμβρίου αναφέρει στην παράγραφο 38 των συμπερασμάτων του ότι απλώ σημειώνει την άποψη τη Επιτροπή για την αίρεση ω προ την έναρξη των διαπραγματεύσεων. Αυτό, κατά την άποψή μου, δεν δηλώνει κατά κανέναν τρόπο αν συμφωνεί με αυτή. Ε, ναι, εγώ επιμένω για τις τροπολογίες αυτές των σοσιαλιστών, αλλά το λέω αυτό στους Έλληνες φίλους μας. Δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν ποτέ τα Σκόπια την έλλειψη συμφωνίας για το όνομα για να μην προχωρήσουν στις μεταρρυθμίσεις. Αλλά κάνω και σε εσά μια έκκληση προς το συμφέρον της χώρας αυτής και προς το συμφέρον της Ευρώπης. Εσείς μην το χρησιμοποιείτε. Το λόγο έχει για ένα λεπτό για την ομάδα των συντηρητικών και μεταρρυθμιστών ο κύριος Τζαμπάσκι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, κύριε Χάν. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να ευχαριστήσουμε τον κύριο Βάικλ για την έκθεση που προετοίμασε και για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει εγώ ως Βούλγαρος και μέλος της ομάδος ECR, υποστηρίζω την ένταξη της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά φυσικά θα πρέπει να εκτιμηθεί αυτή η διαδικασία επί τη βάση των επιτευγμάτων της χώρας αυτής. Η Μακεδονία βρίσκεται σήμερα σε μια κρίση. Έχει υπάρξει υπαναχώρηση από αυτά που είχαν επιτευχθεί στο παρελθόν. Τα μέσα ενημέρωση υφίστανται λογοκρισία. Τα δικαιώματα τη βουλγαρική μειονότητα εκεί παραβιάζονται. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η χώρα αυτή δεν πρέπει να χρησιμοποιήσει το θέμα του ονόματος ως πρόσχημα. Οι αρχές της Μακεδονίας θα πρέπει να προσπαθήσουν να επιλύσουν τα προβλήματα των πολιτών τους, ώστε να έχουν πλήρη δικαιώματα και πλήρης ελευθερίες. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί λοιπόν η ιστορία, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί λόγος πολιτικός που αναμοχλεύει τα μίση θα πρέπει να βοηθήσει να έχει καλύτερες γειτονικές σχέσεις με τους γειτονές της. Τσάνι, you have a blue card. Κύριε Τσάνι, έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα. Γόντα. Ε, köszönöm szépen, tisztelt képviselő úr, ön, mint a szomszédság egyik képviselője. Είστε από γειτονική χώρα, έτσι δεν είναι. Μιλήσατε για τη χώρα αυτή και αναφερθήκατε σε αυτήν ως Μακεδονία και αναφερθήκατε επίσης και στο ζήτημα της ονομασίας. Ξέρετε ότι οι άλλοι χρησιμοποιούν την ονομασία Φιρόμ. Μπορεί η Φιρόμ λοιπόν να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Μακεδονία θα ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα αυτό είναι πολύ σημαντικό και πρέπει να το θεωρώ.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 πολύ καλά ότι ορισμένοι συνάδελφοι δεν το αποδέχονται, θέλουν να λέμε πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία κτλ. Η δική μου πάντω η χώρα έχει αναγνωρίσει την Μακεδονία με την ομασία Μακεδονία. Επομένω αυτό το όνομα χρησιμοποιώ. Σε αυτό το σημείο να μου επιτρέψετε ως προεδρεύων στη συνεδρίαση να αναφερθώ στις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου τις οποίες επανέλαβε για μια ακόμη φορά ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, ο κ. Μάρτιν Σούλτς, με επιστολή του στις 19 Φεβρουαρίου. Σας διαβάζω επιλέξεις στα αγγλικά. Parliament. το Κοινοβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία να χρησιμοποιείται για κάθε ε, σκοπό διπλωματικό και διοικητικό την, ε, το όνομα ΦΥΡΟΜ που είναι το διεθνές αναγνωρισμένο όνομα της χώρας. Λόγο έχει για 1,5 λεπτό η κυρία Σακοράφα. κύριοι συνάδελφοι και με αφορμή την περσινή έκθεση είχα τονίσει ότι η πολιτική της επιτροπής και του κοινοβουλίου να επιβραβεύει την οπισθοδρόμηση όπως παραδεχτήκατε περισσότεροι σήμερα εδώ μέσα και τα αρνητικά αποτελέσματα που συνθέτουν τη σημερινή κατάσταση της χώρας θα λειτουργούσε ανασταλτικά για την πρόοδό της. οι εξελίξεις επιβεβαίωσαν πλήρως το συστημικό έλλειμμα της χώρας σε νευραλγικούς τομείς με αποκορύφωμα την αναβολή των εκλογών του απριλίου ακόμα και σήμερα η ουσία και το περιεχόμενο της πολιτικής συμφωνίας ιουνίου ιουλίου βρίσκεται στον αέρα. τα πολιτικά κριτήρια της κοπενχάγης στα οποία αναφερόμαστε όλοι εδώ μέσα που αφορούν στο κράτος δικαίου στη λειτουργία των δημοκρατικών θεσμών στην ελευθερία έκφρασης στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης και των μέσων ενημέρωσης μόνο αν εθελοτυφλούμε μπορούμε να πούμε ότι πλησιάζουν το ευρωπαϊκό κεκτημένο όσον αφορά δε στο κρίσιμο ζήτημα του προσφυγικού είναι προσβολή να χαρακτηρίζεται το φύρομ ω αξιόπιστο εταίρο όταν καθημερινά παραβιάζει τι διεθνεί συνθήκε με κλειστά σύνορα ποσοστώσει στου πρόσφυγε και περιστατικά βία εναντίον των προσφύγων. πηγαίνετε κύριε συνάδελφοι στην Ιδωμένη για να δείτε πώ συμπεριφέρεται ο αξιόπιστο εταίρο σα. κλείνοντα επαναλαμβάνω το ναυματολογικό δεν είναι διμερέ ζήτημα μεταξύ ελλάδας και φύρομ όπως διατυπώνεται στην έκθεση. είναι διεθνές ανοιχτό ζήτημα και ο μόνος δρόμος για την επίλυσή του είναι η συνέχιση διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του οηε όπως έχουν αποδεχθεί και οι δύο πλευρές η επίλυσή του εντάσσεται αυστηρά στο πλαίσιο των σχέσεων καλής γειτονίας που αποτελούν ουσιώδες στοιχείο της διαδικασίας διεύρυνσης σταθεροποίησης και σύνδεσης και επηρεάζει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα. Κύριοι συνάδελφοι, η ίδια κοντόφθαλμη πολιτική ακολουθείται και με την Τουρκία. Όσο και αν εξυπηρετεί τα συμφέροντα κάποιων, τα αποτελέσματα θα είναι τραγικά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε ευχαριστώ. Για την ομάδα των Πρασίνων τον λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Μέσεριτς. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ο εισηγητής έκανε πάρα πολύ καλή εργασία και με χαρά συνεργάστηκα μαζί του Ο συνήθως το ψήφισμα είναι δυνατό και αξίζει την υποστήριξη όλου του Κοινοβουλίου. Θα μπορούσα να μιλήσω λεπτομερώς για την σημασία της εφαρμογής των συμφωνιών Ιουνίου-Ιουλίου, την ανάγκη των μεταρρυθμίσεων, την ανάγκη όλων των πολιτικών φορέων να αναλάβουν τις ευθύνε τους για να βρουν τρόπους συνεργασίας προς όφελος της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας και προς όφελος του λαού και αυτό θα είναι, είναι αληθές. Αλλά αυτό που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης έχουμε μια ευθύνη στο θέμα αυτό. Δεν είναι μόνο το θέμα του ονόματος. Είναι ένα θέμα, αλλά όχι το μοναδικό. Η σημασία του Συμβουλίου για να βρει μια λύση ευρωπαϊκή στην προσφυγική κρίση είναι ένα από τα στοιχεία που συμβάλλει στην κρίση. Ε, υποσχέσεις ε, του Προέδρου της Επιτροπής για μια περίοδο μεταβατική μετά ε, για περαιτέρω διεύρυνση συμβάλλει ακόμη περισσότερο σε αυτή την κρίση. Πρόκειται για σημαντικές συνεισφορές στην έλλειψη προεπτικές σε όλη την περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων. Χάνουμε, χάνουμε την περιοχή μέρα με την ημέρα και ε, έχουμε μια, ε, ε, ένα, μια ταξία πολιτική. Είναι πάρα πολύ κακή ιδέα. Για την ομάδα Ελευθερίας και Άμεσης Δημοκρατίας, το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κοράου. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Το Μάρτιο του 2004 ξεκίνησε η διαδικασία προσχώρησης της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατία της Μακεδονίας πριν από 12 χρόνια. Σταμάτησε η διαδικασία αυτή και βλέπουμε ότι υπάρχει και μια έντονη αντιπαράθεση ανάμεσα στι πολιτικέ δυνάμει πλέον της χώρα. Εμείς έχουμε το καθήκον να προσπαθήσουμε να επαναφέρουμε την Μακεδονία στο δρόμο αυτό της ένταξης. Και αυτό πρέπει να το κάνουμε βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων, όπως για παράδειγμα μεταρρύθμιση για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ελεύθερα μέσα μαζικής ενημέρωσης, όχι υπό την πίεση της κυβέρνησης. Θα πρέπει να καταπολεμηθεί πραγματικά η διαφθορά σε κάθε επίπεδο. Θα πρέπει να υποστηρίξουμε το δικαστικό σύστημα προκειμένου να μπορεί να λειτουργήσει. Και αυτό προσπαθούμε να δούμε αυτή τη στιγμή και μέσω του ειδικού εισαγγελέα. Να έχουμε τις σωστές κυρώσεις προς τους ενόχους. Αλλά θα πρέπει επίσης να έχουμε και ελεύθερες βουλευτικές εκλογές. Θα πρέπει να έχουμε εκλογικούς καταλόγους οι οποίοι να καταρτιστούν σωστά, προκειμένου οι άνθρωποι να μπορούν ελεύθερα και δίκαια να ψηφίσουν. Έχουμε θέσει λοιπόν κάποιες προϋποθέσεις δημοκρατικές στην Μακεδονία προκειμένου να είναι τελικά μια φιλική χώρα με την οποία θα μπορούμε να συνεργαστούμε. λεπτό για την ομάδα των Εθνών και της Ελευθερίας, ο κύριος Μπέ. Τελικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο οι εκθέσεις επαναλαμβάνονται και μοιάζουν. Και έχουμε δύο απαιτήσει που φαίνονται ότι, ε, από τις οποίες εξαρτώνται ε, η ένταξη κρατών μελών, το ΝΑΤΟ και η προώθηση της ιδεολογίας μας ε, με ε, τις ε, δικές μας διεκδικήσεις. το άρθρο 22 του ψηφίσματος μιλά για το μοντέλο της Ένωσης σχετικά με τις διακρίσεις που οφείλονται στην ταυτότητα του φύλου, ένα, μια αντίληψη ασαφής οι εμμονές σας σας εμποδίζουν να δείτε τα πραγματικά προβλήματα της Μακεδονίας. Μιλάτε για τους Ρωμά. Τι είναι οι τρουβαδούροι που θέλετε να δείτε παντού, εκτός από τους κήπους των δικών σας κατοικιών. Αλλά δεν μιλάτε για τους Αλβανούς της Μακεδονίας, που είναι μια μειονότητα που αυξάνεται δημογραφικά και της οποίας οι διεκδικήσεις απειλούν τη σταθερότητα της χώρας, κυρίως από την ε, δίθεν ανεξαρτησία του Κωσυφοπεδίου. Εκεί υπάρχουν, υπήρξαν από τους Αλβανούς διάφορες διαδηλώσεις, ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους το προσφυγικό και θα ήθελα να επικροτήσω τα μέτρα που έλαβαν οι αρχές της Μακεδονίας στη Σύνοδο Κορυφής των χωρών του Βίζεκράτο ο πρόεδρος έδειξε ότι έχει περισσότερη εμπιστοσύνη στην Ουγγαρία παρά στις Βρυξέλλες για να αναχαιτιστεί η ροή των προσφύγων. ο κύριος Ζαριανόπουλος μία περίπτωση της πρώην ιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας επίσημη ονομασία της χώρας που παραβλέπει η έκθεση στην ευρωπαϊκή ένωση στοχεύει στην ισχυροποίηση του ευρωπαϊκού κεφαλαίου στα βαλκάνια σαν ενεργειακό διάδρομο πεδίο επενδύσεων και γεωστρατηγικό μέτωπο αντιπαράθεσης με τα ρώσικα συμφέροντα. ο λαός της χώρας θα πληρώσει με ακόμα σκληρότερα αντεργατικά μέτρα τα σχέδια της εγχώριας αστικής τάξης. θυμηθείτε η διαδικασία ενσωμάτωσης της φύρομ ξεκίνησε με πόλεμο διάλυση της ιουγκοσλαβίας κράτη προτεκτοράτα του νάτο και της ευρωπαϊκής ένωσης. αποτέλεσμα και της ευρωενωσιακής ενσωμάτωσης της φύρομ είναι το απαράδεκτο κλείσιμο των συνόρων της και του βαλκανικού διαδρόμου στους πρόσφυγες με άγρια αστυνομική καταστολή εγκλωβίζοντάς τους στην ελλάδα για το οποίο η προχθεσινή δήλωση της συνόδου τη συγχαίρει. αυτή η πολιτική που αναπαράγει στο ευρωκοινοβούλιο και η λεγόμενη ομάδα φίλη της μακεδονίας καλλιεργεί εθνοθρησκευτικούς διαχωρισμούς αλυτρωτισμούς αμφισβητήσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων μετατρέποντας τα βαλκάνια κυριολεκτικά σε πυρηνιδαποθήκη. αποδεικνύεται ότι η ευρωπαϊκή ένωση και το σύστημα που υπηρετεί σημαίνουν εκμετάλλευση φτώχεια ανταγωνισμούς και πόλεμο. Σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο Πρέντα. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζουμε όλοι ότι στο τέλος του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν περιέλαβε τη λέξη πρόοδο στην έκθεση για την χώρα αυτή η οποία είναι δυνητικά υποψήφια για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για πολλούς αυτό δεν ήταν καλή επιλογή, αλλά για τη Μακεδονία αυτό ήταν απόλυτα έγκυρο. Δεν μπορεί κανείς να μιλάει για πρόεδρο θα ήταν πολύ καλύτερο να μιλήσουμε για υπαναχώρηση στην περίπτωση της Μακεδονίας, γιατί περί αυτού πρόκειται και η υπεύθυνη για αυτή την κατάσταση είναι η πολιτική τάξη και ιδίω αυτοί οι οποίοι έχουν μποϊκοτάρει το Κοινοβούλιο και έχουν υποστηρίξει την ριζοσπαστική στάση ως πολιτική πρακτική και αυτούς που τους ενθαρρύνουν. Όταν λοιπόν έχουμε μια πολιτική σκηνή όπου το κύριο χαρακτηριστικό είναι η άρνηση του διαλόγου η Μακεδονία βρίσκεται σε μια μόνιμη κατάσταση κρίσης. Για να αλλάξουν τα πράγματα πρέπει όλη η πολιτική τάξη να αντιμετωπίσει με σεβασμό και υπευθυνότητα τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει. Εγώ πραγματικά έχω <clears throat> απογοητευτεί από το πώς οι σοσιαλιστές αρνήθηκαν όλες τις δεσμεύσεις που είχαν αναλάβει έναντι τη διενέργεια των εκλογών που έπρεπε να γίνουν τον Απρίλιο Am văzut că ați lăsat pe toți ceilalți uh, uh, vorbitori să petreacă mult peste timpul alocat. Όλοι οι άλλοι συνάδελφοι και αυτοί ξεπεράσαν το χρόνο που τους είχαν σχεδοθεί. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν με αφήνετε να τελειώσω. Μέσα την απόφαση του Προέδρου που είναι δίκαιος προς όλες τις κατευθύνσεις. Παρακαλώ, καθίστε uh, κάτω. Οι grup. Σεβαστείτε τον Πρόεδρο. Αυτό που κάνετε είναι... Το παραπάνω, μην καταχράσετε την ανεκτικότητά μου. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Νίλσον. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ο κύριος Νίλσον το 2015 μας απέδειξε ότι αντιμετωπίζει τεράστιες προκλήσεις η χώρα αυτή το να καταφέρει τελικά να καταλήξει μια πολιτική συμφωνία, το κυβερνών κόμμα με την αντιπολίτευση, την οποία την είδαμε τον Ιούνιο του 2015, πρέπει αυτή τη στιγμή να δούμε ότι πραγματικά υπάρχει πρόθεση αλλαγή και μεταρρυθμίσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικέ αυτέ για το μέλλον τη χώρα. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι οι ίδιοι οι κάτοικοι τη χώρα να μπορούν να συμμετάσχουν σε δημοκρατικέ εκλογέ. Και δυστυχώ όμω δεν πληρούνται κάποιε βασικέ προποθέσει ακόμα. Για παράδειγμα, ελευθερία των μέσων μαζική ενημέρωση. Χρειαζόμαστε ανεξάρτητα μέσα μαζική ενημέρωση. Αποτελεί αυτό αγοργωνιαίο λίθο οποιασδήποτε δημοκρατική κοινωνία, συμβάλλει σταθερότητα τη χώρα και είναι πάρα πολύ καθοριστικό αυτό για μια ενδεχόμενη προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν όμω εκεί πέρα πολλέ αδυναμίε. Έχουμε έπειτα πολιτική αστάθεια ακόμα στη χώρα, πάρα πολλού μετανάστε οι οποίοι περνάνε από τη χώρα αυτή. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να δείξει μια αλληλεγγύη απέναντι στη Μακεδονία, προκειμένου να αντιμετωπίσει η χώρα αυτή τη σωρία αυτών των προβλημάτων. Η πρόκληση είναι τεράστια. Το πιο σημαντικό όμω είναι να διασφαλίσουμε ότι θα εγκριθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να έχουμε δίκαιε βουλευτικέ εκλογέ. Ένα λεπτό, κύριο Μαριά. Κύριε Πρόεδρε, τα Σκόπια έχουν εδώ και αρκετέ μέρε κλείσει τα σύνορά του με αποτέλεσμα να έχουν εγκλωβιστεί στην Ιδωμένη πάνω από δεκαπέντε χιλιάδες πρόσφυγες. η ενέργεια αυτή των σκοπίων παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και ιδίως τη σύμβαση της γενέβης του 1951 για τους πρόσφυγες όπως άλλωστε δήλωσε και ο γενικός γραμματέας του οηε μπαν Κιμούν. και όμως κύριε χαν δεν είδα να κάνετε καμιά ενέργεια για να αναγκάσετε τα σκόπια να συμμορφωθούν με τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από το διεθνές δίκαιο τα σκόπια επίσης πριν λίγες μέρες παραβίασαν και την εδαφική ακεραιότητα της ελλάδας ρίχνοντας εντός της ελληνικής επικράτειας χειροβομβίδες κρότου λάμψης δακρυγόνα και χημικά προκειμένου να αποθήσουν τους εγκλωβισμένους πρόσφυγες να πλησιάσουν στα σειρματοπλέγματα του έσχους και της ντροπή που έχουν υψώσει. επιπλέον κύριε εισηγητά στην έκθεσή σας πρέπει να χρησιμοποιείτε τον όρο φυρόμ και όχι μακεδονία που κακώς χρησιμοποιείται παραβιάζοντας τις αποφάσεις του οηε που αναγνωρίζουν τα σκόπια με το όνομα φύρομ. δηλώνω κύριε πρόεδρε για άλλη μια φορά ότι είμαι κάθετα αντίθετος σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη ένταξη των σκοπίων στην ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Γιάκοφτσιτς. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω τους συναδέλφους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και να τους συγχαρώ για την εξαιρετική εργασία που κάνουν για την σταθεροποίηση της χώρας αυτής και γενικότερα των Δυτικών Βαλκανίων. Θεωρώ ότι είναι θετικό το ότι προωθούν τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Ελλάδα και θα ήθελα να ενθαρρύνω τους συναδέλφους τόσο στην Ελλάδα όσο και αυτούς που βρίσκονται στην πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας να καταφέρουν να καταλήξουν σε μια πιο συμβαστική προσέγγιση όσον αφορά τα κρεμή ζητήματα. Όσον αφορά την πρωτοβουλία Αδριατική Ιωνίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, πρέπει να σα πω ότι υποστηρίζω το περιεχόμενο τη σχετική έκθεση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταφέρει η Μακεδονία να ενταχθεί στρατηγική Ιωνίου Αδριατικής και μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε έμπρακτα αυτή τη χώρα. Κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν, κάντε παρακαλώ πολύ ό,τι είναι δυνατόν προκειμένου τα 15.000 άτομα τα οποία βρίσκονται στα σύνορα μεταξύ Ελλάδας και Μακεδονίας να καταφέρουν να βοηθηθούν και να επιληθεί βιώσιμα η Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το θέμα της Μακεδονίας έχει οδηγήσει σε μια σειρά από διαμάχες από τότε που διαλύθηκε η Ιουκοσλαβία ως μια χώρα που έχει θέληση να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να γραμμιστεί με την κοινή πολιτική ασφάλεια και εξωτερικών θεμάτων. Εμείς ακούμε συνέχεια ένα επιχείρημα για αυτό να είναι η Μακεδονία μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να χρησιμοποιήσει αυτή την πολιτική μόνο για να υποστηρίξει τα αγγλικά συμφέροντα. Αυτό κατηρικνεί η περίπτωση της Μακεδονίας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν κάνει κάτι υπέρ των κρατών μελών, ακολουθεί μια δική της αυτόνομη λογική που πολλές φορές στρέφεται κατά των κρατών μελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή έχει αντιταχθεί στην αγγλική πολιτική στο Γιβραλτάρ παρά το γεγονός ότι είναι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Ηνωμένο Βασίλειο λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται ούτε και αυτό με θετικό τρόπο και εάν παραμείνουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα συνεχίσουμε να δίνουμε αυτή την άδεια στην Κομισιόν να κάνει τέτοια πράγματα. Έχετε μια μπλε κάρτα από τον κύριο Τάνοκ. Την αποδέχεστε. Κύριε Τάνοκ, έχετε 30 δευτερόλεπτα να θέσετε την ερώτηση. You raised the issue Gibraltar. Μιλήσατε για το Γιβραλτάρ. Δεν είναι θέμα της σημερινή συζήτηση όταν γίνει το Brexit. Τι δυνατότητα θα έχει να ασκήσει πίεση η Αγγλία προς τη Μαδρίτη για να κρατήσει το Γιβραλτάρ ανοιχτό. Γιατί όλοι οι πολίτες του Γιβραλτάρ θέλουν να παραμείνουν στην Ευρώπη και κανείς δεν ψήφισε το κόμμα σας στις τελευταίες εκλογές. Ξέρουν ότι μόνο αν μείνει η Βρετανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορέσει η Ισπανία να κρατήσει ανοιχτό το σύνολο με το Γιβραλτάρ. Παρακαλώ δώστε μου την απάντησή σας. Κύριε Κάρβερ, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Μα κάποια μέρα θα καταλάβετε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι η απάντηση για όλα. Εδώ βρίσκεται η υποκρισία. Υπάρχει ένα κανόνα για τα εδάφη τη Ισπανία στο Μαρόκο και άλλο κανόνα για τα αγγλικά εδάφη στην Ισπανία, το Γιβραλτάρ. Αυτό είναι η υποκρισία. Έχουμε οργανισμούς ε, διεθνείς όπως το Συμβούλιο Ασφαλείας, στους οποίους είμαστε ένα μόνιμο μέλος και θα είμαστε σε πολύ καλύτερη θέση να υπερασπιστούμε τα βρετανικά δικαιώματα και αυτό να περιλαμβάνει και τις ανεξάρτητες επικράτειες παρά να θέλουμε να είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το, αυτήν την αποτυχία της δημοκρατίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συζητάτε αυτά τα θέματα. Περνάμε στον κύριο Επιτίδιο για ένα λεπτό, μία κύριε Πρόεδρε. Το έγγραφο του κυρίου βάγκελ αν και είναι επίσημο έγγραφο, αναφέρει σε πολλές περιπτώσεις την ε, λέξη Μασεντόνιαν κατά παράβαση της διοντολογίας προκαλώντας ταυτόχρονα και την ε, ελληνική ευαισθησία πάνω στο θέμα αυτό. Γι' αυτό θα έπρεπε αυτό να αποφευθεί. Κατά τα άλλα, αποκαλύπτει ε, τα ελλείμματα δημοκρατίας που υπάρχουν στα Σκόπια. Τα πολιτικά κόμματα δεν μπορούν να συμφωνήσουν για τη διεξαγωγή των εκλογών και αναβάλουν συνεχώ την ημερομηνία τη διεξαγωγή. όμω ακόμη και αν ε, διεξαχθούν αυτέ οι εκλογέ ουδή γνωρίζει εάν θα διεξαχθούν με δημοκρατικέ διαδικασίε και αν τα αποτελέσματά του θα είναι αποδεκτά. επίση στη χώρα επικρατεί διαφθορά δεν υπάρχει ελευθερία τύπου δεν υπάρχει ανεξαρτησία τη δικαιοσύνη παρεμποδίζεται το έργο του ειδικού εισαγγελέα ε, ο ρόλο του κοινοβουλίου είναι περιορισμένο και παραβιάζονται τα δημοκρατικά δικαιώματα παράλληλα τα σκόπια παραβιάζοντας την υποχρέωση μιας υποένταξη χώρας ε, να δημιουργήσει συνθήκες καλής γειτονίας προκαλούν την ελλάδα κλείνοντας τα σύνορά της. μετά λοιπόν την κλοπή της ιστορίας του πολιτισμού αλλά και την έκφραση και τη διατύπωση επεκτατικών ε, βλέψεων κατά της ελλάδος έχουμε και το κλείσιμο των συνόρων. με αυτή την προβληματική χώρα θέλετε να διεξάγουμε ενταξιακές συνομιλίες. δεν μας φτάνει η τουρκία. θέλουμε να εκθρέψουμε και άλλον εκβιαστή. Διερωτώ με σε αγεντικά κλιμάκια της ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πολιτικός μαζοχισμός. ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κούκαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθου καρδία τον κύριο Βάκλη για την εκθέσή του. Η Μακεδονία βρίσκεται σε μια δύσκολη κατάσταση. Η πολιτική κρίση δεν έχει ξεπεραστεί και μαζί με τις μεταναστευτικές ροές δημιουργούν μια ιδιαίτερα εύθραυστη κατάσταση στη χώρα αυτή. Εγώ πιστεύω ότι η χώρα αυτή χρειάζεται την υποστήριξή μας. Η διαδικασία ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κλειδί για το μέλλον της χώρας αυτής. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τις προσπάθειες και να βοηθήσουμε τη χώρα αυτή να ενισχύσει την πολιτική σταθερότητα και τη δημοκρατία. Για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε θα πρέπει να υπάρξει πλήρη συμφωνία της πολιτικής συμφωνίας του προηγούμενου έτους και επομένως αμερόληπτες και ελεύθερες εκλογές τον Ιούνιο και εφαρμογή των κατεπηγουσών προτεραιοτήτων για μεταρρύθμιση. Είναι κρίμα που η Μακεδονία εξακολουθεί να περιμένει την, το άνοιγμα των διαπραγματεύσεων για 7 πια χρόνια και τώρα ενώπιον αυτών των προκλήσεων θα πρέπει να διπλασιάσει τις προσπάθειές της για να κινηθεί στον δρόμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να τη βοηθήσουμε. Ευχαριστώ. έχει για ένα λεπτό κύριος Πιτσούλα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. prijepori oko imena bez konkretnog napretka ali se s druge strane nažalost politička situacija u zemlji postupno pogoršavala. zato i pozdravljam dogovor vlasti i oporbe Είμαστε. Ωραία, μηδενίζουμε το χρόνο παρακαλώ και ξεκινήστε από την αρχή κύριε Πιτσούλα και ζητώ συγγνώμη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχά τον κύριο Βάιγκλ γιατί κάνει ένα πολύ αντικειμενικό απολογισμό ενό πολύ δύσκολου έτου για την ε, ΦΥΡΟΜ του έτους 2015. Γίνονται αυτή τη στιγμή κάποιες συστάσεις προκειμένου να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις. Έχουμε πει ότι δεν έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ με το ζήτημα της ονομασίας. Παράλληλα όμως ε, διαβρώνεται η κατάσταση πολιτική στη χώρα. Είμαι σαφώ λοιπόν υπέρ τη συμφωνία τη Πρίστινα, η οποία μπορεί να συμβάλλει πάρα πολύ στην πολιτική συμφωλήση στην χώρα αυτή. Διαφορετικά τα προβλήματα θα γίνουν χρόνια προβλήματα και ενδεχομένω να επηρεάσουν και τι γύρω περιοχέ. Θα πρέπει να βοηθήσουμε όλου ιδιαίτερω στη Μακεδονία αυτή τη στιγμή, ακριβώ επειδή πλήττεται ω χώρα διέλευση από την μεταναστευτική κρίση. Επίση υπάρχουν πολλά εσωτερικά προβλήματα σε ένα περιβάλλον γεωπολιτικό το οποίο είναι ιδιαίτερα εύθραυστο. Είχαμε κάποια εσωτερικά φαινόμενα όπως οι υποκλοπές τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, φαινόμενα διαφθοράς. Όλα αυτά έχουν οδηγήσει σε βαθιά ρήγματα στην κοινωνία και σε έλλειψη πολιτικού διαλόγου. Αν λοιπόν καθυστερήσουν ακόμα περισσότερο μεταρρυθμίσεις, πολύ φοβάμαι ότι θα μειωθεί ακόμα περισσότερο η εμπιστοσύνη των πολιτών. Χριστοφόρου, έχετε 30 δευτερόλεπτα για το ερώτημα παρακολουθώ τη συζήτηση κύριε πρόεδρε και θλίβομαι πραγματικά που το ευρωκοινοβούλιο που ουσιαστικά κίδεται της δημοκρατίας και της νοημότητα και αντί να σεβαστεί τις αποφάσεις του οργανισμού ηνωμένων εθνών όσον αφορά την ονοματολογία των σκοπίων επιμένουν κάποιοι συνάδελφοι αντί του σωστού ονόματος φύρων να αναφέρονται σε μακεδονία. αυτό που δεν κατόρθωσε ο τίτο μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο που ουσιαστικά δημιούργησε έτσι θελικά ένα νέο έθνος και μοίρασε τα ελληνικά σύμβολα και την ελληνική ονομασία προσπαθούμε εμεί ω ευρωκοινοβούλιο ανιστόρητα να επιβάλλουμε έτσι θελικά ένα όνομα που είναι καθαρά ελληνικό η μακεδονία είναι ελληνικό πολιτισμό, ελληνική ονομασία ελληνική ιστορία θέλουμε έτσι θελικά να το επιβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο να δικαιώσουμε τον τίτο που δεν τα κατάφερε αυτό όταν προσπαθούσε να το επιβάλλει. Είναι σαφέ το ερώτημα. Κύριε Πιτσούλα, έχετε 30 δευτερόλεπτα για την απάντηση. Αγαπητέ συνάδελφε, καταλαβαίνω απόλυτα τις ευαισθησίες σας όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Οφείλω όμως να σας πω ότι στα πλαίσια του διεθνούς διαλόγου η Μακεδονία αναγνωρίζεται με το όνομα το οποίο φέρει στο Σύνταγμά της αλλά και με το όνομα το οποίο χρησιμοποιείτε εσείς, το Φύρομ δηλαδή. Η δική μου η χώρα, η Κροατία, έχει αναγνωρίσει τη Μακεδονία βάσει του σταγματικού της ονόματος. Ανεξάρτητα από τις δικές ευαισθησίες, εμείς θα χρησιμοποιούμε και στο μέλλον το όνομα αυτό και ελπίζουμε ότι η Σκόπια και η Αθήνα θα καταλήξουν σε συμφωνία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, κυρίε και κύριοι. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Βάικλ για τη θαυμάσια έκθεσή του. Επίσης εκτιμώ αυτό το οποίο έχει κάνει και ο κύριος Χάν σε σχέση με την βραδία διαδικασία αυτή. Φυσικά δεν υπάρχει καμιά άλλη δυνατότητα διαδικασίας διεύθυνση τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ είμαι υπέρ αυτή τη διαδικασίας και πιστεύω ότι η Μακεδονία ή η Φιρόμ, αν θέλετε να χρησιμοποιήσω αυτό το όνομα, πρέπει να θεωρηθεί τμήμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και για να το πω πιο ουδέτερα η θέση των Σκοπίων είναι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεν θα ήθελα τα προβλήματα εσωτερικής δημοκρατίας στη χώρα αυτή να χρησιμοποιηθούν ως πρόσχημα για την καθυστέρηση της πορείας της χώρας αυτής προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω ότι οι προσπάθειες αυτής της χώρας να προχωρήσουν να Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι. Εγώ πιστεύω ότι τρία σημεία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει η Φιρόμ να επανέλθει στη σωστή τροχιά. Καταρχήν όλες οι πολιτικές δυνάμεις πρέπει να υπομισθούν τις ευθύνες τους και να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή των δεσμεύσεών τους με βιώσιμο τρόπο. Δεύτερον, η χώρα πρέπει να ετοιμαστεί για τις κοινοβουλευτικές εκλογές και να εξασφαλίσει την αμερόληπτη διαδικασία στις εκλογές. Τρίτον, ο αγώνας κατά τη διαφθορά πρέπει να συνεχιστεί με αποφασιστικό τρόπο. Η πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας χρειάζεται την υποστήριξή μας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι το ψήφισμά μας θα συμβάλλει σημαντικά στο να διατηρηθεί η χώρα στην ευρωπαϊκή της πορεία και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Ιβο τον εισηγητή. Ναι. Ένα λεπτό, ο κύριος Φρουντζουλίτσα. Κυρίες και κύριοι, σημειώνω την απόφαση του Κοινοβουλίου της Μακεδονίας 23 Φεβρουαρίου να ορίσει νέα ημερομηνία για πρόορες εκλογές την 16 Ιουνίου. Το γεγονός ότι δεν υπήρχε κονσένσου στην αντιπολίτευση είναι κάτι το λυπηρό και είναι μια χαμένη ευκαιρία. Οι μεταρρυθμίσεις στα μέσα δεν μπορούν να γίνουν παρά μόνο μετά τις εκλογές όλα τα πολιτικά κόμματα στην Μακεδονία πρέπει να καταβάλουν προσπάθειες για να δημιουργήσουν τις συνθήκες για τις πρόορες εκλογές και κάθε ε, συμφωνία είναι πάρα πολύ ε, σημαντική βάση της ε, Συμφωνίας Πριτζίνα. Η πρόοδος των προτεραιοτήτων πρέπει να συνεχιστεί η Ελλάδα και η Βουλγαρία δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για να παρεμποδίζεται η διαδικασία ενταξιακή στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά να χρησιμοποιούνται επικοδομητικά το νωρίτερο δυνατόν στην διαδικασία λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές των Ηνωμένων Εθνών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Την Σπυράκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχετε το λόγο για 30 δευτερόλεπτα αν θέσετε το ερώτημά σας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε συνάδελφε, σας άκουσα προσεκτικά να μιλάτε για διμερεί ζητήματα και διαφορές στην περιοχή. Ωστόσο θα ήθελα να σας θέσω υπόψη το εξή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Οργανισμού Δημοσιογράφη Χωρίς Σύνορα που αξιολογεί την ελευθερία του τύπου, η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας κατατάσσεται στη θέση 117, 90 θέσεις χαμηλότερα από ό,τι βρισκόταν το 2009 είναι η τελευταία στην ευρώπη. υπάρχουν σοβαρότατες τρευλώσεις στην νομοθεσία στην έκφραση των μέσων ενημέρωσης στην παρέμβαση από το κράτος μέσω διαφήμισης. θα ήθελα να σας ρωτήσω δεν σας απασχολεί η παραβίαση ενός τόσο σοβαρού κριτηρίου στην καρδιά της ευρωπαϊκής ένωσης για μια χώρα που ζητά ημερομηνία ένταξης; Κύριε Φρουντσούλητσα, έχετε 30 δευτερόλεπτα με τη σχετική ανοχή, όσοι έδειξα και στην κυρία Σπυράκη. Uh, Η Μακεδονία θα πρέπει να συμμορφωθεί με όλα τα προαπαιτούμενα, όλα αυτά τα θέματα πρέπει να τα επιλύσει. Αυτό είναι σαφέ. Αλλά συγχρόνω δεν μπορούμε να αφήσουμε όλε τι χώρε των Δυτικών Βαλκανίων σε μια φαιά περιοχή. Είναι απαραίτητο σιγά σιγά να ενσωματώσουμε όλε αυτέ τι χώρε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ, αν θέλουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον αυτού του φορέα που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι σημαντικό για όλου μα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Τάνοκ. Μακεδονία είναι μία μικρή χώρα, δεν έχει πρόσβαση στη θάλασσα, αντιμετωπίζει πάρα πολλές εντάσεις στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό η χώρα αυτή να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να καταφέρει τελικά να προεδρεύσει, προκειμένου να καταφέρει να βελτιώσει την οικονομία τη. Πρέπει να υποστηρίξουμε λοιπόν την υποψηφιότητα τη χώρα αυτή, ζητώντα από τα κράτη-μέλη που έχουν εκκρεμεί ζητήματα αυτή τη στιγμή να καταλήξουν σε κάποιε λύσει, ιδίω όσον αφορά το ζήτημα τη ονομασία. Στα πλαίσια τη πενταστατική κρίση, ξέρετε ότι η Μακεδονία αντιμετωπίζει πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Έρχονται επίση και εκλογέ τον Ιούνιο. Όλα αυτά τα ζητήματα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα, ιδίω όσον αφορά την, τις ιδιαίτερες σχέσεις που είχαμε με τη χώρα αυτή και την κατάσταση της χώρας που είναι ιδιαίτερα εύθραυστη. Για πάρα πολύ καιρό έχουν σταματήσει οι ταξιακές διαπραγματεύσεις. Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, γιατί ούτω ή άλλω θα ακολουθήσουν αρκετά χρόνια μέχρι να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθότι προωθούνται περισσότερο οι όμορε χώρε τη, δεν θα ήθελα να φτάσουμε σε ένα σημείο που τελικά η Μακεδονία θα είναι απλώ μία υποψήφια χώρα, περιτριγιζόμενη από χώρε που θα έχουν ήδη ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ πριν από αυτήν. Κύριο Πλένκοβιτς, τη δέχεστε. Κύριε Πλένκοβιτς, έχετε 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Τάνοκ, είπατε ότι υποστηρίζετε την προσχώρηση της Μακεδονίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την έναρξη των διαπραγματεύσεων ένταξης αν λάβουμε υπόψη την έκθεσή σας για το Μαυροβούνιο και τη συμμετοχή της χώρας αυτής στο ΝΑΤΟ, θεωρείτε ότι η Κομισιόν έχει δώσει αρκετά χρήματα για να ξεπεραστεί η δύσκολη κατάσταση στα σύνορα μεταξύ Μακεδονίας και Ελλάδος στην κατάσταση αυτή η οποία κλιμακώνεται συνέχεια. Αυτό δεν έχει άμεση σχέση με το Μαυροβούνιο για το οποίο είμαι εισηγητής. Το Μαυροβούνιο δεν έχει συνοριακές πιέσεις όπως οι Μακεδονίες. Εγώ νομίζω ότι κάπου 700 εκατομμύρια έχουν δοθεί, δεν θυμάμαι ακριβώς, έχουν δοθεί ως βοήθεια και προφανώς η Μακεδονία βρίσκεται σε τεράστια πίεση με το κλείσιμο των συνόρων αλλά πιστεύω ότι δεν μπορεί κανείς να έχει απεριόριστους αριθμούς μεταναστών. θα πρέπει να υπάρξει μια συμφωνία. Είδαμε τη συμφωνία που έγινε με την Τουρκία και ελπίζουμε τώρα ότι αυτή θα είναι αποτελεσματική για να μειωθεί η ροή προσφύγων. Ελπίζω ότι τα Δυτικά Βαλκάνια θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση και το πρόγραμμα με την Τουρκία θα δώσει στους ανθρώπους τη δυνατότητα να παραμείνουν στους καταβλισμούς τους στο Λίβανο, την Ιορδανία και την Τουρκία και όχι στην Ευρώπη μέσω των Βαλκανίων. Το λόγο έχει για ένα λεπτό ο κύριος Κεφαλογιάννης πρόεδρε το πρόβλημα για τις διαπραγματεύσεις ευρωπαϊκής ένωσης σκοπίων δεν είναι το όνομα είναι το έλλειμμα δημοκρατίας που υπάρχει στην πρώην ιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας. κύριε πρόεδρε ο σεβασμός στα κριτήρια της Κομπεχάγης είναι το ζητούμενο και στα κριτήρια της κοπεχάγης συμπεριλαμβάνονται και ο σεβασμός των σχέσεων καλής γειτονίας μεταξύ των κρατών στην έκθεση της ευρωπαϊκής επιτροπής έχει υπογραμμιστεί η οπισθοδρόμηση στα θέματα δικαιοσύνης στα θέματα διαφάνειας στα θέματα της λειτουργίας των μέσων μαζικής ενημέρωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος. η χρησιμοποίηση από, ε, την έκθεση του επιθέτου μακεδονικός ουσιαστικά δίνει την αίσθηση ότι το ευρωπαϊκό κοινοβούλιο λαμβάνει θέση υπέρ των σκοπίων το ζήτημα της ονομασίας δεν είναι ζήτημα διμερές είναι ζήτημα διεθνές και ως διεθνές ζήτημα πρέπει να λυθεί μέσα στα πλαίσια του οργανισμού των ηνωμένων εθνών. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει για 1,5 λεπτό ο κύριος Βάιντεν Χόλτσερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφερθήκαμε σε πάρα πολλά προβλήματα όπως η ε, διαφθορά, Υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις ε, οι οποίες μπορούν να εξηγηθούν ε, με τις ελλείψεις της χώρας. Η μεγαλύτερη πρόκληση για τη χώρα είναι αναμφίβολα η προσφυγική κρίση. Σχεδόν όλοι οι πρόσφυγες ε, ταξιδεύουν μέσα από τη χώρα αυτή για να πάνε στην Ευρώπη. Τα Σκόπια αντιμετώπισαν αυτή την πρόκληση ακόμα και με βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τώρα, κατά πόσον τηρήθηκαν οι ευρωπαϊκές προδιαγραφές, τα ευρωπαϊκά κριτήρια, αυτό δεν μπορούμε να το πούμε. Και μιλάω από προσωπική εμπειρία. Έχω πολλές φορές διανύσει τη Βαλκανική Οδό. Ε, βεβαίως πρέπει να πούμε ότι οι πολίτες βοηθούν, οι ΜΚΟ και οι εθελοντές ε, προσπαθούν να προσφέρουν περίθαλψη και νομική αρρωγή. Από την άλλη υπάρχουν ε, εκθέσεις που δείχνουν ότι υπάρχουν πάρα πολλοί διακινητές και την τελευταία τελευταία φορά στη Γευγελή ε, διαπίστωσα μόνιμος μου ότι ε, ασκείται και βία έναντι των προσφύγων. Τέτοιου είδους ε, καταστάσεις καταλαβαίνετε ότι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το πόσο έτοιμη είναι η χώρα να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά θα πρέπει να προβληματιστούν και εκείνοι οι οποίοι νομίζουν ότι η χώρα αυτή... Ένα λεπτό, κύριος Πέτερλε. Eh, Ευχαριστώ για την υπεύθυνη εργασία του και για την απάντηση σε θέματα. Η πολιτική εξέλιξη πέρσι ε, θα μας έδειξε ότι η ευρωπαϊκή πρόπτικη της Μακεδονίας, της ΦΥΡΟΜ, δεν εξαρτάται μόνο από την βούληση και από τις μεταρρυθμίσεις και την Ευρώπη, αλλά και από την εσωτερική σταθερότητα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Λυπούμε που οι συνέπειες των εσωτερικών εξελίξεων για πρώτη φορά είναι ένας όρος ε, στις συστάσεις και στα σχόλια και γιατί μόνο η ε, συνεπής εφαρμογή μπορεί να αυξήσει την αξιοπιστία της ενταξιακής διαδικασίας και να σταθεροποιήσει ε, την εικόνα αυτής της υποψήφιας χώρας. Και θα ήθελα να τονίσω την πρόοδο που έχει γίνει στην περιοχή για την Ευρωπαϊκή Τροχιά. Κύριε Πρόεδρε, η ευρωπαϊκή οικοδόμηση δεν μπορεί να είναι πλήρης χωρίς τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θα μιλήσουμε για την μετανάστευση, αλλά υπάρχουν άλλα προβλήματα παλαιότερα και βεβαίως ό,τι υποδαβλίζει το μίσος δεν πρέπει να είναι μέρος. Όσοι ε, θεωρούνται ότι είναι φίλοι στην Βουλγαρία ε, δεν πρέπει να λαμβάνονται υποτάσεις, έχουν επαναληφθεί πολλές φορές και διαρωτώ ε, γιατί υπάρχει όλη αυτή η δυσπιστία ε, από την κομμουνιστική εποχή ε, και δεν έχει ξεπεραστεί και έχουμε τον Πίταν ο, ο οποίος μου είπε ότι δύο βιβλία του παππού του έχουν δημοσιευθεί στα Σκόπια παραβιάζοντας τους κανόνες και αναφέρονται ως Μακεδονία και Η Βουλγαρία έχει αντικατασταθεί με τη λέξη Μακεδονία. Αν η Μακεδονία θέλει πράγματι να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τις δύσκολες σημερινές συνθήκες, στον δρόμο προς την Ευρώπη θα πρέπει να υπερνικήσει αυτά τα σφάλματα του παρελθόντος. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βάικλ για την έκθεσή του και τον ευχαριστώ γιατί δέχτηκε μερικέ από τι τροπολογίε μου για την ε, προσχώρηση τη Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ και τι ενταξιακέ διαπραγματεύσει με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ ότι η χώρα αυτή έκανε τη μεγαλύτερη πρόοδο στι ενταξιακέ διαπραγματεύσει και στην ευθυγράμμιση με το κοινοτικό κεκτημένο. Γι' αυτό είναι άδικο να την κρατάμε 10 χρόνια στον προθάλαμο, στην αίθουσα της Ε, Θα ήθελα λοιπόν να ε, καλέσω το Συμβούλιο να επιληθούν ε, γρήγορα τα και τα διμερή θέματα. Ε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα των εκλογών στη Μακεδονία. Θεωρώ ότι θα πρέπει να μην ε, παίξουμε το παιχνίδι αυτών που θέλουν να, να, δια, να κυβερνήσουν χωρίς εκλογές. Ε, φυσικά χρειάζονται μεταρρυθμίσεις, αλλά η Μακεδονία έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο στη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης, γιατί γι' αυτό και χρειάζεται ισχυρότερη υποστήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Μακεδονία χρειάζεται την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση τη Μακεδονία. Γι' αυτό ζητώ από το Συμβούλιο να ξεκινήσει ε, διαπραγματεύσει με τη Μακεδονία, λέει ο Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να συγχαρώ τον κύριο Βάιγκλ για την έκθεσή του και να ήθελα να πω και να απευθύνω δύο εκκλήσεις προς τον Επίτροπο της Διεύρυνσης, τον κύριο Χάν. Θα πρέπει καταρχήν να ενισχύσουμε τις διοικητικές ικανότητες αντιπροσωπείας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία έχασε 70 εκατομμύρια ευρώ ε, από τα κονδύλια που δικαιούνταν. Θα πρέπει να έχουμε μια κεντρική διαχείριση αυτών των ε, ε, χάρη στην ενίσχυση των διοικητικών ικανοτήτων της αντιπροσωπεία μας. Δεύτερη έκκληση αφορά την επιστροφή των 70 εκατομμυρίων ευρώ προ τη Μακεδονία ώστε να αξιοποιηθούν για τη διαχείριση τη μεταναστευτική κρίση. γιατί η χώρα αυτή ε, καταβάλει μεγάλε προσπάθειες για τη διαχείριση των συνόρων και την ε, σωστή υποδοχή των μεταναστών. Γιατί το να χάνει μια μικρή χώρα 70 εκατομμύρια είναι μεγάλο ποσό. Γι' αυτό σα παρακαλώ να λάβουμε υπόψη ότι ε, αυτά που κάνουμε για τη Μακεδονία θα πρέπει ε, να τα εφαρμόσουμε και αυτά που είχαμε εφαρμόσει με άλλες χώρες που ήταν συνταξιακή διαδικασία θα πρέπει να επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις. Γραμμένων ομιλητών για την έκθεση προόδου 2015 για την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Περνάμε στην διαδικασία Catch the Eye. Έχω δεχτεί οκτώ αιτήματα από σχεδόν όλες τις πολιτικές ομάδες. Θα τα δεκτώ όλα. Παρακαλώ να είστε συνεπείς στο χρόνο που είναι ένα λεπτό. Η κυρία Σουλίν Πατρίτσι έχει το λόγο για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να συγχαρώ τον συνάδελφο τον κύριο Βάγκλ για την εξωτερική του έκθεση. Υπό αυτές τις περιστάσεις όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει προβλήματα με την προσφυγική κρίση, η Μακεδονία, λέει μιλήτρια, απέδειξε ότι είναι πολύ αξιόπιστος εταίρος. Παρά την δύσκολη εσωτερική πολιτική κατάσταση που αντιμετωπίζει και παρά τις επικείμενες εκλογές η χώρα αυτή τήρησε τους κανόνες του Σέγγεν πολύ περισσότερο από τις χώρες μέλη του χώρου Σέγγεν. Φαίνεται βέβαια ότι οι ανακοινώσει τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ίδιε από χρόνο σε, χώρο, ή χρόνο σε χρόνο. Η Μακεδονία όμω είναι έτοιμη και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λοιπόν θα πρέπει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξεκινήσει διαπραγματεύσει με τη Μακεδονία. Καπούτ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ανησυχούμε πάρα πολύ για την κατάσταση στη ΦΥΡΟΜ. Εκεί αφορά τα δικαιώματα και τι θεμελιώδει ελευθερίε. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχουν ακόμα πολλέ ε, διεθνωτικέ εντάσει ε, και δεν βοηθάει αυτή η προσέγγιση για του πρόσφυγε. Ε, εκατομμύρια ή χιλιάδε, αν θέλετε, έχουν στριμωχτεί στα σύνορα με την Ελλάδα και αφήνουν να περνάνε μόνο πολύ λίγοι μετανάστες, ε, εκείνοι οι οποίοι έχουν έγγραφα από την Ελλάδα. Τα Σκόπια έχουν ε, την ανάγκη της Ευρώπης, αλλά είναι σημαντικό να ευθυγραμμιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η διαδικασία είναι δύσκολη, πρόκειται για χώρες οι οποίες δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα τις δικές τους τις πολιτικές επιλογές. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Επίτροπε, κύριε Χάν, είχα πει πριν από ένα χρόνο ότι η ένταξη των Βαλκανικών χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεμελιώδη σημασία και αυτό θα πρέπει να γίνει χάρη τη κοινωνία των πολιτών. Δυστυχώ ε, η Μακεδονία έχει μείνει πίσω. Αυτό μπορεί να θέσει ένα αμφιβόλο την ενταξιακή πορεία αυτή τη χώρα. Είναι μία από τις ε, χώρες που ανήκουν στη λεγόμενη Βαλκανική Οδό, η Βαλκανική Διαδρομή των προσφύγων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ανοίξει τους κόλπους της και προς τη χώρα αυτή και να ξεκινήσει τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Έτσι θα στηρίξουμε την ενταξιακή πορεία, την ευρωπαϊκή πορεία αυτής της χώρας. Επίσης θα πρέπει οι εκλογές να τηρούν τις διεθνείς προδιαγραφές. Και ας μην ξεχνούμε ότι δεν θα πρέπει να μελούμε τις μειονότητες στη Μακεδονία. Μόνο έτσι θα επιστρέψει η εμπιστοσύνη στους θεσμικούς φορείς και θα γίνουν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας των Σκοπίων κατά το έτος 2015 είναι αποκαλυπτική. Δέκα ολόκληρα χρόνια μετά την απόκτηση του καθεστώτος της υποψήφιας για ένταξη χώρας δεν έχει γίνει καμία πρόοδος στο θέμα της ονομασίας και στην αποκήρυξη των εδαφικών διεκδικήσεων κατά της ελλάδας τις οποίες υποκρύπτει η ονομασία. αντίθετα οι σχέσεις καλής γειτονίας επιβαρύνονται από την πλαστογράφηση και το σφετερισμό της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και με την ανέγερση αλόκοτων μνημείων στην πόλη των σκοπίων πέρα από αυτά υπάρχει οπισθοδρόμηση σε κρίσιμους τομείς όπως είναι η εμπέδωση της δημοκρατίας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα με το καθεστώς Γκρούευσκι να κινείται σε ολοένα πιο αυταρχική κατεύθυνση. σε κανένα από τα θέματα αυτά δεν μπορούν να γίνουν εκπτώσεις εκ μέρους της ευρωπαϊκής ένωσης και επομένως δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων. σας ευχαριστώ. Το λόγο έχει επίσης για ένα λεπτό ο κύριος Σόλτες. Σας ε, ευχαριστώ πάρα πολύ ε, αγαπητέ συνάδελφε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ε, ενέργεια και το δυναμισμό που επενδύσατε σε αυτή την έκθεση που είναι εξαιρετική. Η Μακεδονία βρίσκεται στον προθάλαμο για πάνω από δέκα χρόνια και η Μακεδονία βρίσκεται σε μια ιδιαίτερη θέση όσον αφορά τη συμμετοχή της σε σύγκριση με άλλες χώρες των Δυτικών Βαλκανίων που είναι επίσης υποψήφιες. Βεβαίως η Μακεδονία εξακολουθεί να αντιμετωπίζει πολλές προκλήσεις αλλά η κρίση το, το προσφυγικό είναι πολύ σημαντική κρίση και η Μακεδονία απέδειξε ότι είναι σε θέση να φέρει ένα μεγάλο βάρος παρότι είναι μικρή χώρα. Θεωρώ λοιπόν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αντί να μιλά και να αναλώνεται σε λόγια θα πρέπει να δράσει. Εξάλλου και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αντιμετωπίσει τη Μακεδονία κάτω από διαφορετικό πρίσμα γιατί από τη μια ε, παραβλέπουμε αυτά που κάνει η Τουρκία όχι όμως αυτά που κάνει η Μακεδονία. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι τον συνάδελφο κύριο Βάγγελ για την πάρα πολύ καλή δουλειά που έκανε με την έκθεσή του που ο συνήθως είναι μια έκθεση ειλικρινής, ισορροπημένη η οποία δείχνει ότι έχουν γίνει βήματα προς τα εμπρός αλλά υπάρχουν ακόμα πολλές ελλείψεις η κυβέρνηση ΦΥΡΟΜ μεταρρυθμίσεις που πρέπει να προχωρήσουν με μεγαλύτερη συνέπεια όσον αφορά τη δικαιοσύνη που είναι ακόμα επιλεκτική, ε, τον, ε, τη δημόσια δημόσια διοίκηση, τη διαφθορά, τα προβλήματα τα διεθνωτικά και ακόμα περισσότερο την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης. Εμείς είμαστε πεπισμένοι ότι πράγματι θα πρέπει να υπάρξει διεύνηση για όλες τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων. Θεωρώ όμω ότι θα ήταν ε, ολέθριο λάθος αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο να ε, χορηγήσουν ενταξιακό καθιστώ στη Μακεδονία. Ε, δεν είναι δυνατόν η χώρα αυτή να παίζει τον ρόλο του τροχονόμου και η Ελλάδα, ίσως αργότερα και η να γίνουν αποθήκες ψυχών σε σχέση πάντα με τον μεταναστευτικό. Αυτό είναι ένα λάθος. Εμείς θέλουμε διαδικασίες ελεύθερες και ισορροπημένες για τη Μακεδονία. Για ένα λεπτό η κυρία Σπυράκη. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριοι συνάδελφοι κύριε Χάν, το ερώτημα είναι τι ζητάμε από τις υποψήφιες για ένταξη χώρες συμμόρφωση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο με τα κριτήρια της κοπενχάγης. τι συμβαίνει στην πρώην γιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας; έχει σοβαρό έλλειμμα στο διαχωρισμό των εξουσιών στο σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων στο σεβασμό της ελευθερίας του τύπου είναι τελευταία στην ευρώπη ενενήντα θέσεις κάτω από το. δύο χιλιάδες θα ανοίξουμε σήμερα το δρόμο των εκπτώσεων και πώς θα απαντήσουμε έτσι στις απαιτήσεις της τουρκίας σε όσα καταγράφουν οι πρέσβεις της ευρωπαϊκής ένωσης και των ηνωμένων πολιτειών που οδήγησαν στην αναβολή των εκλογών προστίθεται και η συμπεριφορά της πρώην γιουγκοσλαβικής δημοκρατίας της μακεδονίας σήμερα στα ελληνοσκοπιανά σύνορα εκεί όπου δεν επιτρέπεται να περάσουν πρόσφυγες που χρήζουν διεθνούς προστασίας. συνάδει αυτό με το πνεύμα και το γράμμα των ευρωπαϊκών αποφάσεων; η πρώην ιουγκοσλαβική δημοκρατία της μακεδονίας έχει ακόμη πολύ δρόμο να διανύσει να λειτουργήσει η δημοκρατία της όπως οι ευρωπαϊκές δημοκρατίες και τότε να ανοίξουμε την πόρτα της ευρωπαϊκής ένωσης. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει για ένα λεπτό και με αυτόν κλείνουμε τη διαδικασία του Catch ο κύριος Πόλτσακ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν θα ήθελα να υπάρχουν εκκρεμότητες που να μπλοκάρουν την ενταξιακή πορεία της χώρας αυτής. Ε, δυστυχώς έχουμε μείνει πίσω στις μεταρρυθμίσεις στη ΦΥΡΟΜ. Ε, θα πρέπει να πραγματοποιήσει πρώτα τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις η χώρα αυτή και μετά να περιμένει την πλήρη υποστήριξή μας στην ενταξιακή της πορεία. Οι ανησυχίες που εξέφρασαν οι συνάδελφοι είναι εύλογες. Ε, είναι αναφυσβήτητο ότι η ΦΥΡΟΜ χρειάζεται τη βοήθειά μας, αλλά θα πρέπει να κάνει και τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Είμαι μάλιστα και μέλος της ομάδας φίλη τη ΦΥΡΟΜ. Το λόγο έχει ο Επίτροπος κ. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη, σας ευχαριστώ πάλι και άλλη μια φορά για τη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρίως εκείνους που ε, παρέμειναν μέχρι το τέλος, παρακολούθησαν όλη τη συζήτηση. Πιστεύω ότι οι πολιτικοί ηγέτες ε, της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας φέρουν πλέον την ευθύνη να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε η χώρα να επανέλθει στην Ευρωατλαντική Οδό. Εκπέμψαμε ένα σαφές μήνυμα ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει πολιτική συμφωνία, ε, να εφαρμοστούν επιγόντω οι μεταρρυθμίσει. Εξάλλου, η χώρα έχει δεσμευτεί προ αυτή την κατεύθυνση. Η πρόκληση που αντιμετωπίζουν οι πολιτικοί ηγέτε είναι να επιδείξουν πολιτική βούληση και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε στι 5 Ιουνίου να λάβουν χώρα ε, ανώθευτες και αδιάβλητες εκλογές αυτό είναι σημαντικό στη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων. Οι εκλογές πρέπει να επαναφέρουν την εμπιστοσύνη των πολιτών στη χώρα, στην κυβέρνηση. Με τη δική σας λοιπόν την υποστήριξη θα συνεχίσουμε ε, στην κατεύθυνση που έχουμε χαράξει. Θα παρακολουθούμε εκ του σύναγκη στη χώρα. Η χώρα δεν έχει καιρό να χάσει και αυτό το λέω και σε σχέση με αυτά που αναφέρθηκαν εδώ επανειλημμένα. Προφανώς εννοώ το μεταναστευτικό, τις προσφυγικές ροές. Πιστεύω λοιπόν ότι η πολιτική ηγεσία της ε, χώρας πρέπει να εστιάσει την προσοχή της σε αυτά τα προβλήματα. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει τη χώρα με τεχνογνωσία, με χρηματοδότηση, αλλά ε, θέλω πάλι να επαναλάβω ότι όλα αυτά γίνονται μετά από αξιολόγηση. Δεν είναι ότι εκταμιεύουμε κονδύλια έτσι γενικά και αόριστα, παρά μόνο εφόσον υπάρχει ε, ανάγκη ε, η οποία μπορεί κάπως και να στηριχθεί. Η πολιτική λοιπόν κρίση πρέπει να τελειώσει και αυτό είναι προς όφελος της χώρας. Θέλω να ελπίζω είναι προς όφελος ε, και των πολιτών. Υπολογίζω λοιπόν σε εσά, στην υποστήριξή σας για να στείλουμε ένα ενωμένο μήνυμα στην πολιτική ηγεσία αυτής της χώρας και σε όλους εκείνους οι οποίοι επέκριναν τις δημοκρατικές εξελίξεις στη χώρα αυτή να σας πω επιτρέψτε μου ότι η κριτική που ασκήσατε είναι δικαιολογημένη, συμφωνώ μαζί σας. Από την άλλη βέβαια οφείλουμε να καταλάβουμε ότι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, για τα δικά μας τα συμφέροντα, το σημαντικότερο όλων είναι να έχουμε διαπραγματεύσεις όπου θα μπορούμε να επισημάνουμε αυτές τις ελλείψεις. Μόχλευση των ετοιμάτων μας μπορεί να προκύψει μόνο μέσα από τη συζήτηση και επίσης και κατά τη διάρκεια των ε, διαπραγματεύσεων. Ε, υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα όπου μετά στο ε, πέρας των συζητήσεων δεν έχουμε δυνατότητα άσκησης επιρροής. Μιλάμε για την ε, περαιτέρω εξέλιξη της ε, πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Θέλω να προσβλέπω στην υποστήριξή σας και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ όχι μόνο για τη σημερινή συζήτηση αλλά γενικότερα για τη στράτευση που επιδεικνύεται. Το λόγο έχει η κυρία Χένης Πλασάρτ και πρώην συνάδελφός μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, αξιότιμοι ευρωβουλευτέ. Θα ήθελα εν κατακλείδη να εκφράσω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη προς τον εισηγητή τον κύριο Βάγκλ, αλλά και προς κύριο Χόλτ και Κούκαν για την πολύ αξιόλογη προσπάθειά τους. Το Συμβούλιο αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη πρόοδου με την πρώην Ιουκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Βέβαια, είμαστε και θα παραμείνουμε ιδιαίτερα ανήσυχοι ως προς την έθραυστη χώρια πολιτική κατάσταση. Η ανάγκη επικοδομητικού διαλόγου αφορά όλους τους παράγοντες του, της πολιτικής σκηνής και όλους τους βασικούς πολιτικούς εταίρους. Η σύσταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων πάγεται στην πλήρη υλοποίηση των συμφωνιών του Ιουνίου και την σημαντική πρόοδο στις πεταρρυθμίσεις ε, που θα πρέπει να γίνουν κατά προτεραιότητα. Και αυτό είναι σωστό. Ε, θα δούμε το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών και μετά θα σας ενημερώσουμε για τη συζήτηση στο Συμβούλιο. Τώρα του στους ηγέτες της πρώην Ιουκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας να δείξουν αποτελέσματα και χαίρομαι που οι περισσότεροι συμφωνήσατε ως προς την προσέγγιση αυτή. Περιμένουμε τη συνεχή συνεργασία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και υπολογίζουμε σε αυτήν ώστε να καλέσουμε όλου του ηγέτε των πολιτικών παρατάξεων τη πρώην Οικοσλαβική Δημοκρατία τη Μακεδονία για καλόπιστη συνεργασία προκειμένου να επανέλθει η χώρα στον, στη μεταρρυθμιστική τη πορεία. Αυτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε έλαβα μία πρόταση ψηφίσματος για την περάτωση αυτής της συζήτησης. Η συζήτηση έληξε. Η ψηφοφορία θα